του θέματος αυτού και θα ακολουθήσει αργότερα η ψηφοφορία. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ειδικότερη περίπτωση δύο κρατουμένων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Ιβ Μακβαμπάλα και του Φρέντ Μπάουμα. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στους συντάκτες των ψηφισμάτων. Πρώτη θα λάβει το λόγο η κυρία Σαρτζεντίνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο που παραμείνατε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει την προσοχή για να δούμε τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι. Ο Μακ Παμπάλα και ο Φρέντ Μπάουμα που είναι φυλακισμένοι στην Κισάσα του συνέλαβαν ε, ως ηγέτες ε, μιας οργάνωσης νεολαίας που διαδήλωνε για περισσότερη δημοκρατία και κατά του νέου εκλογικού νόμου στο Κονγκό. Φιλίμπι λέγεται αυτό το κίνημα και προσπαθεί να βελτιώσει τη δημοκρατία στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και πατάσετε και καταστέλετε βία. Εμείς λοιπόν ζητούμε από το Κοινοβούλιο να αφαιθούν αμέσα ελεύθεροι η Ιβ Μακ Βαμπάλα και ο Φρέντ Μπάουμα γιατί ε, είναι ακτιβιστές δημοκράτες και στην Κινσάσα και στην Κόμα ε, ε, εκδηλώθηκαν κινήματα αλληλεγγύης. Εκτός αυτού ζητούμε να δοθεί προσοχή και σε ένα μαζικό τάφο που ε, ανακαλύφθηκε κοντά στην Κινσάσα τον Απρίλιο ε, που είναι γεμάτο ε, λείψανα, ανώνυμα, δεν ξέρουμε σε ποιους ανήκουν, αγνοούμενοι και η κυβέρνηση στην Κινσάσα λέει καλά δεν τρέχει και τίποτα. Η οργάνωση Human Rights Watch το έχει ερευνήσει και λέει ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι ε, σωρή ακτιβιστών που θέλει να ξεφορτωθεί η κυβέρνηση. Ε, ε, εμείς θέλουμε να υποστηριχθούν οι αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί και της δημοκρατίας και καλούμε την κυβέρνηση της χώρας να ε, το διερευνήσει αυτό εξονυχιστικά και καλούμε και τις οικογένειες των αγνοωμένων να κινητοποιηθούν και να ενημερωθούν από την κυβέρνηση για ε, την τύχη των αγαπημένων τους. Φέτος γίνονται εκλογές, είναι προεκλογική χρονιά ε, στο Κονγκό και κινδυνεύει η κατάσταση να εκτροχιαστεί. Εμείς θα πρέπει να παρακολουθούμε τι συμβαίνει γιατί θα ήταν τρομακτικό να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Αυτό που εμείς ζητούμε είναι να υπάρχει ένα μέλλον για τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρα. Ε, Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κοράο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η κατάσταση που συζητάμε τώρα για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ε, μοιάζει πολύ με αυτή ε, που συζητήσαμε για τον Μπουρούντι. Ε, κρατούμενοι ακτιβιστές που φυλακίζονται επειδή εκφράζουν αντίθεση προς την κυβέρνηση, προς τη βούληση του Προέδρου να ανανεώνει επαόριστον την κυβερνητική θητεία, εξαφανίζονται ή καταλήγουν στη φυλακή και είναι σαφές ότι με αυτό το ψήφισμα εμείς εκφράζουμε την υποστήριξή μας προς αυτούς τους ακτιβιστές και ζητάμε από την κυβέρνηση της Κινσάσα να ελευθερώσει αμέσως αυτά τα δύο παιδιά που φυλακίστηκαν. Όσον αφορά τη λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο, πιστεύω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε τις δεσμεύσεις της στην κυβέρνηση στο πλαίσιο των συμφωνιών της Κοτονού. Πρέπει να σεβαστούν και να τηρήσουν αυτές τις συμφωνίες και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πραγματοποιηθεί αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δεμεσμάκερ, παρακαλώ. Ε, ε, στο Μπουρούντι και στην κεντρική, κεντροαυτοκανική δημοκρατία ε, είναι ταραγμένα τα πνεύματα και τώρα και στο Κονγκό και νέοι ε, Κονγκολέζοι θέλουν να παίξουν ρόλο για να βελτιώσουν τη ζωή της χώρας τους. Πριν από τρεις μήνες ξεκίνησε μια πρωτοβουλία των νέων που ε, κατεστάλλει και ε, συνελήφθησαν 30. Οι περισσότεροι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι αλλά διοργανωτές Μακφαμπάλα και Μπάουμα ε, κρατούνται ακόμα και είναι ύποπτοι εθνική προδοσία. Είναι τεράστιο το πρόβλημα ταυτότητας που έχει η χώρα. Από τη μια έχει πάρα πολλούς νέους με τεράστιο ταλέντο και από την άλλη προσκρούν όλα αυτά ε, σε μια ε, διεφθαρμένη κυβέρνηση. Το νοσοκομείο στο Μπάνζι του δόκτωρα Μοκφέγε ε, Μοχάβε έχει ε, τελείως ε, ε, παράλογα κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή και για πλήρωτους λογαριασμούς. Και ο δόκτωρ Μουγουάμπε είναι εκείνος που γνωρίζετε ότι τιμήθηκε πέρσι με το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δημοκρατική, ε, λέει, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, μόνο δημοκρατία δεν είναι. Τι ηρωνία είναι αυτή. Βέντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το κοινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο είναι ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα προς τις αρχές της χώρας. Γι' αυτό, όπως και άλλοι, και εγώ ζητώ την άμεση απελευθέρωση του Φρέντ Μπάουμα και του Ιβ Μακβαμπάλα από το νεανικό κίνημα του Φιλίμπη στο Κονγκό. Είναι ηρωνία το ότι έχει μπροστά ε, την... Ε, ε, λέξη λαϊκή δημοκρατία η χώρα αυτή όταν βλέπουμε τέτοιες έντονες αντιδράσεις από πλευράς των αρχών Επίσης, ό,τι αφορά ε, τις ε, αρχές της νεολαίας, ε, δεν μπορούν να δεχθούν περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης των δικαιωμάτων του συνεταιρίζεστε. Έχασαν τη ζωή τους στο Γενάρη τουλάχιστον 12 διαδηλωτές. Αυτό δείχνει ότι βγαίνει εκτός ελέγχου η κατάσταση για τις αρχές της Κινσάσα και αντίστοιχα γεγονότα βλέπουμε στον Μπουρούντι. Σε ένα χρόνο περίπου θα γίνουν εκλογές στο Κονγκό. Η στήριξη εκλογική διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα στη βασιστεί στο κατά πόσον οι συστάσει ε, τη παρατή εκλογών θα υλοποιηθούν. Ευχαριστώ. Μαρή Κριστίν Βερζιά για 1,5 λεπτό τώρα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ για τα καλά σας γαλλικά, κύριε Πρόεδρε. 25 χρόνια δικτατορίας, 15 χρόνια εμφυλίου αναρχιστρωμένου από τις γειτονικέ χώρες που θέλουν να ελέγξουν ιδίω το εξορρυκτικό πλούτο και με βάση την κάρτα 7 εκατομμύρια νεκροί. Έχουμε παράνομη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου που έχει να κάνει με δισεκατομμύρια μόνο για στην ανατολική χώρα. Έχουμε επίσης ε, διεθνή εγκληματικότητα. Πρόκειται για μια χώρα που ε, χυμάζεται. Κάποιοι έχουν πληρώσει με τη ζωή τους, όπως ο Φλωρίμπε Σαμπαγιά. Έχουμε βίες αματηρές ε, καταστολές, όπως ε, τον Ιανουάριο. Γιατί ο Ζωζεύ Καμπιλά θέλει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο να μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία. Κυρίω οι ακτιβιστέ κοινωνία των πολιτών είναι στόχοι. Η νεολαία, το κίνημα Φιλίμπη και επίση πολλοί προσφυγέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιβ Μακουβαμπάλα και ο Φρέτ Μπάουμα είναι σύμβολα που ζητούν ε, την ε, απελευθέρωσή τους ε, και 15 ΜΚΟ και 20 και οργανώσεις ζητούν το ίδιο. Πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την απελευθέρωση και όπως ζητάει η αντιπολίτευση να συμμετάσχουμε και σε μια διεθνή προσπάθεια διαμεσολάβησης για να έχουμε έναν διαφανή διάλογο που θα συμμετέχουν όλοι πριν τι τελευταίες, πριν τις επόμενες εκλογές. Νομίζω ότι το δικαιούται αυτό ο λαός του Κονγκό. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Νάρτ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ και εγώ για τα ωραία σας ισπανικά, πρόεδρε. Το να τη λένε λαϊκή δημοκρατία είναι οξύμορον, είναι εσωτερική αντίφαση. Δυναστεία είναι που βασίζεται στη διαφθορά και στην καταστολή. Και υπόθηκαν ήδη, λέγοντας αυτά, τα έχουμε πει όλα. Θα μπω αμέσως στην ουσία. Κοιτάξτε, η Ευρώπη μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Να ασκήσει τη δημοκρατική υποκρισία, δηλαδή άρθρο 2, δημοκρατική ρήτρα στις συμφωνίες που ποτέ δεν την εφαρμόζουμε και έχουμε τη συμφωνία Κοτονού με το άρθρο 8, 9 και 96 που σε ελάχιστε ευκαιρίε έχουν υλοποιηθεί. Αν είναι λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό θα πρέπει να τη στείλουμε ένα μήνυμα κατηγορηματικό και ξεκάθαρο. Τι να το κάνουμε το ψήφισμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μια τρύπα στο νερό. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το σημείο 13 και παρακαλώ να το έχετε υπόψη σας. Να απαιτήσουμε όντως να επιδείξουν την αντίστοιχη συμπεριφορά με το σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου κτλ και έχει αναλάβει αυτές τις δεσμεύσεις η χώρα και αν δεν εφαρμοστεί ε, κατά τρόπο ριζοσπαστικό και απόλυτο ε, τότε θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα άρθρα 9 και 96. Τι να τα κάνουμε τα ψηφίσματα, γιατί βαφκαλιζόμαστε. Εδώ πρόκειται για δημοκρατική υποκρισία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βάιτενχολτσε. Ένα λεπτό. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό είναι μια χώρα γεμάτη αστάθεια, παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καθημερινή υπόθεση και μας απασχολεί συχνά η χώρα εδώ. Τελευταία φορά το Μάιο όταν πρόκειται για τα ορυκτά ε, από εμπόλεμες περιοχές και πέρσι όταν ο δόκτωρ Μουκβέγγε πήρε το βραβείο Ζαχάροφ. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή η γιορτή αυτή και μας εξήγησε πώς έχει η κατάσταση στη χώρα και πώς έχουν οι συσχετισμοί. Απευθύνθηκε στο θεωρείο προς τους μετανάστες από το Κονγκό που ζουν εδώ, οι οποίοι τον επεφημούσα και είπε ε, ότι η χώρα ε, θα πρέπει να αλλάξει τώρα που βρισκόμαστε. Έχουν συλληφθεί οι δύο ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι αυτοί και πολλοί άλλοι. Απαιτούμε να φεθούν ελεύθεροι και απαιτούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαντλήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της και τις πιέσεις που μπορεί να ασκήσει, έτσι ώστε ε, του χρόνου μετά τις εκλογές του 2016 να μπορέσει να βρει μια ειρηνική πορεία η χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουλευτά. Pitches on behalf of groups. First of all, Τώρα η ομιλία για τις ομάδες, ε, των ομάδων. Πρώτος εκ μέρους του Έλκε η κυρία Μαρία Αρένα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ήθελα απλά να διακρίνησω ότι είμαι από τους σοσιαλιστές κύριε Πρόεδρε. Ζητά συγγνώμη ο Πρόεδρος, κανείς δεν είναι τέλειος, λέει. Νομίζω το ΕΛΚ δεν θα το ήθελε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Φρέντ Μπομά και ο Ιβ Μακουαμπαλά είναι δύο νέοι πολίτες ε, του Κονγκό που αυτή τη στιγμή κρατούνται στην Κισάνσα απλά και μόνο διότι συναντήθηκαν με άλλους νέους ε, Αφρικανούς, με άλλα κινήματα της Αφρικής για να αγωνιστούν για τα ε, δικαιώματα του πολίτη, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Αυτοί οι δύο νέοι βρίσκονται τώρα φλεξμένοι στο Μακαλά μετά από μερικούς μήνες ε, στα κρατητήρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και η δίκη έχει μόλις ξεκινήσει ε, σήμερα όπου κατηγορούνται ότι επιχείρησαν ε, κατά τη ζωή του Προέδρου απλά γιατί συναντήθηκαν και εμείς απαιτούμε ως Ευρώπη την άμεση φυλάκισή τους και θέλουμε επίσης να ζητήσουμε από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να ακυρώσει όλες τις κατηγορίες προς αυτούς όπως και προς τα κινήματα Φιλιμπή και Λουτσά διότι τα κινήματα αυτά είναι σημαντικά στη σημερινή προεκλογική εκστρατεία που είναι τεταμένη και ε, αυτό το κίνημα θα πρέπει να ε, ε, δώσει κάποια δημοκρατικά δικαιώματα στους νέους του Κονγκό οι οποίοι πρέπει να αγωνιστούν για την ελευθερία και την δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ζητώ και πάλι συγγνώμη. Είστε εκπρόσωπος φυσικά των σοσιαλιστών. Επόμενος ομιλητής, ε, η, ε, η κυρία Χαράντσοβα από το Άλντε. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών είναι ζωτική σημασία για οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία. Στο Κονγκό η ε, οι οργανισμοί κοινωνίας των πολιτών ε, συμπληρώνουν το ρόλο ενός κράτους που δεν παρέχει ε, ό,τι χρειάζονται οι πολίτες του. Οι ειρηνικοί συναντήσεις δεν μπορούν να τιμωρούνται. Δεν μπορεί το Κονγκό να απαγορεύει στο λαό του να συναντάται και να κινητοποιείται. Το ότι στοχεύονται κινήματα νέων και πολιτικοί αντιφρονούντες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ως πρώτο βήμα για τη συμφιλίωση με το δικό του λαό ο, ε, ο, ε, τον το, πρέπει να ελευθερωθούν ο Ιβ Μακβαμπαλά και ο Φρέντ Μπάουμα και όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι επίσης πρέπει η χώρα να χρησιμοποιήσει όλα τα ωφέλη και να τα που, τα ωφέλη που προσφέρει μια δυναμική κοινωνία των πολιτών η οποία όχι απλά ελέγχει το κράτος αλλά προσφέρει και στην κοινωνία τη δυνατότητα να επιλύει κοινά προβλήματα. Έχει έρθει η ώρα οι αρχές του Κονγκό να το δουν αυτό ως προνόμιο και όχι ως απειλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Κατσδιάε. Α, το συγγνώμη. Κατσδιάε. Ο κύριος Βανέκοφτσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν είναι η αρχή της εκλογικής, ε, προεκλογικής εκστρατείας ή ε, οι δύο άνθρωποι αυτοί είναι ε, τα σύμβολα ε, της ε, αντίστασης και τι θα γίνει. Το θέμα είναι ποιος θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται αυτή τη χώρα και να ωφελείται από τα όσα συμβαίνουν στο Κονγκό. Χωρίς πολιτισμό, χωρίς δημοκρατία. Ποιος στην Ευρώπη είναι η ερώτηση, ωφελείται. Ποιος έχει συμφέρον ε, να ισχύει αυτό το καθεστώς στο Κονγκό και να παραμένει αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα γιατί έχει συμφέροντα η Ευρώπη στη χώρα αυτή, στο Κονγκό και αν τα έχει θα πρέπει να βοηθήσουμε τη φιλική αυτή χώρα να βάλει τα του οίκου της εντάξει. Μάξιμο, Μάσιμο Καστάλτο τώρα. Ευχαριστώ. Στη γλώσσα σας κύριε Πρόεδρε ο Ιβ Μακουαμπάλα και ο Φρεντ Μπάουμα. Ο αγώνας του είναι και δικό μας. Διαφορετικά συναδελφέ λυπάμαι. Δεν έχει νόημα να, δίνουμε, να πονέμε το βραβείο Σαχάροφ και μετά να το ξεχνάμε. Είναι η επέτειος ε, της γενοκτονίας στη Ρουάντα και ακόμα στις χώρε ε, χώρες ε, έχουμε πολέμους. Αυτοί οι δύο ε, άνθρωποι φυλακίστηκαν γιατί υπερασπίστηκαν την ελευθερία της ε, συνάντησης. Βρέθηκαν ένα σωρό νεκροί μέσα σε ε, ομαδικούς τάφους και υπάρχουν ίσως και άλλοι αντιφρονούντες όπως είπε ο συνάδελφος Νατ πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να τηρούνται οι συμφωνίες του Κοτονού και όλες οι υπόλοιπες. Εγώ θέλω εδώ να αντιχήσουν τα λόγια του Φρεντ Μπάμ όταν είπε ότι δεν θα δεχτούμε ποτέ ε, το, η διαδρομή ε, ελευθερίας και δημοκρατίας ε, να παρεμποδίζεται από κάποιους. Θα υπερασπιστούμε την δημοκρατία στη χώρα μας, την έλευση της δημοκρατίας και κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει, ούτε οι αυθαίρετες συλλήψεις. Ας μην αφήσουμε να πεθάνουν οι δημοκρατικές φιλοδοξίες της νεολαίας του Κονγκό. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, κάποιος Ευρωβουλευτή. Κύριε Πρόεδρε, εσείς αστειάκια κάνετε, λέτε τους σοσιαλιστές εδώ, ΕΛΚ. Ε, κάποιοι γέλασαν, το θεώρησαν ανέκδοτο, καθόλου ανέκδοτο δεν είναι. Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στο ΕΛΚ και στους σοσιαλιστές. Γιατί για να διατηρήσουν το status quo τα έχουν κάνει πλακάκια παρασκηνιακά στο Κοινοβούλιο και όλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κονγκό. Ενώ κοιτάξτε τι γίνεται στην Ουγγαρία. Το 2006 υπήρξε βίαιη καταστολή από πλευρά τη αστυνομία με φυλακίσει κατά δεκάδε πολιτών σε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, θυμίζω τότε στην Ουγγαρία κυβερνούσαν. Ε, και τώρα ε, κυβερνάει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο λογοδοτεί αστυνομία και και που προσπαθούν να προστατεύσουν τους πρώην σοσιαλιστές συναδέλφους. Οπότε καμία διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μόρβαη. Now, uh, on behalf... Και τώρα εξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο έχει η Επίτροπος η κυρία Μάλστον. Παρακαλώ. Thank you very ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται πράγματι για μια πολύ σοβαρή συζήτηση και πρέπει να σας ε, διαβεβαιώσω ότι ακούσαμε τα πολύ ξεκάθαρα μηνύματά σας και θα διαβιβάσουμε και στην υπάτη εκπρόσωπο. Θεωρούμε ότι η Ολομέλεια μας δίνει στήριξη για να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης ε, της υποθέσεις του κύριου Μακουαμπάλα, του κυρίου Μπάουμε και όλων των υπολείπων. 30 άτομα έχουν ε, στην Κινσάσα συλληφθεί φέτος ε, στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου που είχε οργανώσει το κίνημα Φιλίμπη. Προσπαθεί να ε, κινηθεί με πολύ υπεύθυνο αστικό τρόπο. Υπήρξαν κάποιοι οποίοι απελευθερώθηκαν ή ε, απελάθηκαν. Είναι δύο όμως ε, ακόμη στις φυλακές και πάνω από 40 μέρες κρατούνταν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών χωρίς ε, δυνατότητα νομικής υπεράσπισης. Πήγαν στο γραφείο της Αγγελέα όπου τους απαγγέλθηκαν διάφορες κατηγορίες. Μιλάμε για αυτά τα δύο άτομα τον Ιβ Μακβαμπάλα και τον Φρέντ Μπάουμα. Πολύ λίγε πληροφορίε έχουμε στη διάθεσή μα. Φαίνεται όμω ότι είναι αβάσιμε, αστήρικτε οι καταγγελίε αυτέ και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ μεγάλο ο κίνδυνο να είναι πολιτική λόγοι της κράτησής τους. Πρέπει να απελευθερωθούν οι δύο αυτοί κρατούμενοι γιατί με την κοινοβουλευτική έρευνα δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο ότι οι ηγέτες ή συμμετέχοντες σε αυτό το εργαστήριο Φιλίμπη είχαν ε, σκοπό να προγραμματίσουν τρομοκρατικές επιθέσεις ή βίες ενέργειες. Οι ηγέτες ε, όμως γι' αυτό κατηγορούνται, για το ε, Φιλίμπη, συγκεκριμένα για πρόκληση βίας εξέγερσης και προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων. Δεν υπάρχει όμως τίποτα που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Είναι κενέ αυτέ οι καταγγέλίε. Εμεί συνεχίζουμε να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά αυτέ τι ε, ε, υποθέσει. Έχουμε κάνει διαβήματα δύο φορέ ο Υπουργό Δικαιοσύνη ε, και υπάρχουν και, και παρατήρησαν την δικαστική διαδικασία. Μπορείτε να βασιστείτε στο ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Τώρα, γενικότερα, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λέτε ότι πρέπει να είναι στο επίκεντρο του διάλογο που έχουμε με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που έχει πολυμορφία απόψεων, κομμάτων, φιλοδοξιών και πάνω απ' όλα φέτο είναι σημαντικό οι πολιτικοί φορεί, οι αστικοί φορεί να μπορούν να μιλούν ελεύθερα ε, και να μπορούν να δημοσιοποιούν τις απόψεις τους, ε, να γίνεται διάλογο. Ο σεβασμό στο διάλογο, στα ανθρώπινα δικαιώματα σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό σκέλο τη Συμφωνία του Κοτονού και είναι και σημαντικά ζητήματα και τον εκλογικό κύκλο που ξεκινά από τώρα μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. Θέλουμε να στηρίξουμε τη διαδικασία αυτή. Πρέπει να υπάρχουν όμως οι προποθέσει προϋποθέσεις ότι αφορά χρονοδιάγραμμα, πολιτικό κλίμα και προπολογισμό και στις τοπικές δηλώσεις και στα συμβούλια, ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου εκφράζουμε τις ανησυχίες μας ε, ε, γιατί περιορίζεται το πολιτικό φάσμα ιδίως με την αναθεώρηση του νομοσχεδίου για το εκλογικού νόμου στις αρχές του έτους. Θα μπορούσε να υπάρξει ενορχίστρωση, χειραγώγηση ή να εξπετήσει πολιτικές σκοπιμότητες κάτι τέτοιο και να οδηγήσει σε προσαγωγές, συλλήψεις, αυθαίρετες κρατήσεις, αχρίαστη χρήση βίας, φυσικών απειλών και εκφοβισμού φοβισμού των δημοσιογράφων. Όταν τα μέλη ε, της υπηρεσία πληροφοριών ε, κάνουν παράνομες ενέργειες θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα έρευνα ε, και δίωξη. Έχουμε τον Αφρικανικό χάρτη για τη δημοκρατία, τις εκλογές, τη κυβέρνηση και τονίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ανοιχτό διάλογος, να προστατεύεται η ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα της αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρχει αμεροληψία και ανεξαρτησία. Εμείς θα στηρίξουμε ε, σε μια γνήσια εταιρική σχέση το η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, έχουμε ε, και τη δέσμευση των 620 εκατομμυρίων. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να μιλάμε, να υψώνουμε τη φωνή μας όταν έχουμε ανησυχίες, όπως στην προηγουμένη περίπτωση, αλλά και σε πολλές άλλες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στη γλώσσα σας, τάκ, σας ευχαριστώ στα Σουηδικά. Ε, Ευχαριστώ πολύ και στα πολωνικά τώρα. Λοιπόν, προχωρούμε. Έχω λάβει 7 ε, προτάσεις ψηφίσματος ε, από τις συνήθεις πολιτικές ομάδες της